πραγματικά καλοσύνη σας που αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά πραγματικά σήμερα εμείς πενθούμε. Ευχαριστώ κυρία Δεκεζέρ και νομίζω ότι όλοι είναι στο πλευρό σας αυτή την οδύνη και σας συμπαρίστατε. εκφράστε παρακαλώ την αλληλεγγύη ε, στα θύματα. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση που είχαμε και περνούμε αμέσως στην επόμενη που αφορά τη δήλωση της Αντιπροέδρου της ε, Πάτης Εκπροσώπου για ε, την ε, Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Σας δίνω αμέσως το λόγο κυρία Άστον χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ δια της κυρίας Δεκεζέρ να διαβιβάσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό το γεγονός στη Λιέγη. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωση Ρωσία, που όπω γνωρίζετε ε, αρχίζει αύριο το βράδυ στις Βρυξέλλες. Ε, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια και για τι εκλογέ προηγουμένω, όπω γνωρίζουν τα μέλη, κοινοβουλευτικέ εκλογέ για την κρατική δούμα έγιναν στη Ρωσία στι 4 Δεκεμβρίου. Όταν τον Ιούλιο εδώ συζητούσαμε την προετοιμασία των εκλογών αυτό, εξέφρασα κάποιε ανησυχίε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό στην πολιτική πολυφωνία. Στη συνέχεια, μετά από αυτές τις παρατηρήσεις σήμερα, η εκ των προτέρων ε, εξαίρεση και αποκλεισμό ορισμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης ε, επηρέασε αρνητικά τις εκλογές. Επίσης είδαμε ε, προβλήματα στη διαδικασία όπως η μεροληψία των μέσων ενημέρωσης και επίσης συμμετοχή του κόμματος ε, στην εξουσία σε κάποιες ε, δράσεις. Ε, ανησυχούμε για την κράτηση και σύλληψη και κράτηση διαδηλωτών και ακτιβιστών καθώς και δημοσιογράφων. Καλωσορίζω τις εντολές που έδωσε ο πρόεδρος Μετβέτεφ έτσι ώστε να ε, διερευνηθούν όλες οι κατηγορίες. Ε, η εκλογική νομοθεσία στη Ρωσία προβλέπει και ένσταση και επανόρθωση και περιμένουμε να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Θα πρέπει να μελετηθούν αυτά και ο ΑΣΕΙ, και άλλοι οργανισμοί εν ευθέτω χρόνο θα ε, εξάγουν τα συμπεράσματα σε εκθέσεις. Θα πρέπει να γίνει αυτό έτσι ώστε να είναι ομαλές και ταχύες Προεδρικέ εκλογέ το Μάρτιο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο ρωσικός λαός έκανε χρήση όλων των δυνατοτήτων που είχε να εκφράσει και τη δυσφορία του προς ε, ορισμένε καταστάσει σήμερα. Πολλοί ε, σχολιαστές λέγουν ότι οι ε, ψηφοφόροι εξέφρασαν την άποψή τους απέναντι ε, στη διαφθορά, την έλλειψη πολιτικών ελευθεριών και την οικονομική κατάσταση ψηφίζοντας άλλα κόμματα. Οπότε το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας από το 64% που είχε πάρει το 2007 είναι κάτω από το 50% σήμερα. Οι Ρώσοι πολίτες έστειλαν ένα μήνυμα σαφές που σίγουρα ελήφθη και ο πρόεδρος ε, Μετβέντεφ και ο πρωθυπουργός Πούτιν έλαβαν το μήνυμα. Οι των δημοκρατικών θεσμό στη Ρωσία, όπω είπα τον Ιούλιο, θα εξαρτηθούν από το ρωσικό λαό και τι επιλογέ του. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν είναι ε, απαθείς παρατηρητής. Έχουμε κοινούς δεσμούς οικονομικούς και κοινή ιστορία. Ως στρατηγική εταίρεια από κοινού μπορούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία να αντιμετωπίσουν ε, προκλήσεις και να ασκήσουν σημαντική επιρροή παγκοσμίω. Επίσης έχουμε αναλάβει κοινέ δεσμεύσει για να αναπτύξουμε δημοκρατικούς θεσμούς στα πλαίσια του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. Βεβαίω, ε, θα θέσουμε υπόψη των αρμοδίων αύριο τι ανησυχίε μας. Για, για εμάς ε, ξεχρονισμό σημαίνει ε, ένταξη της Ρωσίας στο σύστημα των διεθνών κανόνων και ενίσχυση των ελευθεριών των πολιτών. Πραγματικά η σύνοδος Κορυφή μπορεί να οδηγήσει σε πολλά αποτελέσματα, λειτουργεί η συνεργασία. Ε, ε, επιτρέψτε μου καταρχάς να μιλήσω για την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ που κανονικά επισήμω θα εγκριθεί ε, στη Γενέβη την Παρασκευή. 18 χρόνια διήρξαν διαπραγματεύσεις και ήταν σημαντικός εταίρος η Ρωσία. Ως πρώην Επίτροπος Εμπορίου είχα και ίδια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα είναι ιστορική στιγμή που θα σημάνει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Θα συνδέσει τη Ρωσία στους διεθνείς εμπορικούς ε, κανόνες, θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για εμπόριο και επενδύσεις και θα προστατεύσει τις δικές μας εταιρείε από αυθαίρετες αποφάσεις. Θα δοθεί λοιπόν νέα όθηση και στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση Ρωσία. Για τη θεώρηση διαβατηρίων και την κινητικότητα, οι πρόεδροι θα εγκρίνουν ένα κατάλογο κοινών ε, βημάτων προς ε, ταξίδια χωρίς θεωρήσει. Η διαδικασία άρση θεωρήσεων σημαίνει σημαντικό εξυγχρονισμό σε τομεί όπω είναι η διαχείριση συνόρων και οι πολιτικέ μετανάστευση αλλά και ο σεβασμό των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η βελτίωση κινητικότητα και οι επαφέ των ανθρώπων μεταξύ του θα βοηθήσουν στην ανταλλαγή εμπειριών, αξιών, ε, στην πολιτιστική συνεργασία και στι επιχειρήσει. Επίσης, η εταιρική σχέση για εξυγχρονισμό είναι σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή με νέα προγράμματα. Στη Σύνοδο Κορυφής θα διατρανώσουμε και πάλι την πεποίθησή μας ότι ο εξυγχρονισμός δεν σημαίνει τεχνολογία και μόνο. Κράτος δικαίου, προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, κοινωνία των πολιτών και ίση κανόνες βεχνιδιού για όλες τις εταιρείε είναι κρίσιμα στοιχεία για μια επιτυχημένη διαδικασία εξυγχρονισμού. Ε, Τελειώντα, να πω δύο λόγια για την εξωτερική πολιτική. Είναι σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ρωσία. Ε, με τον Σεργέη Λαυρόφ συνεργαζόμαστε τακτικά. Γενικά επιτυχάνουμε, αλλά σε κάποιε περιπτώσει δίστανται οι απόψει μα. Το προφανέ παράδειγμα τη εποχή είναι η που σίγουρα θα συζητηθεί και στις συνοδοκορυφής. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, και στις παγωμένες σειράξεις στην υπερδριστερία. Ε, καταφέραμε να ξεκινήσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις 5 συν 2. Χρειάζεται ε, υποστήριξη και για το Ρινό Καραμπάχ, ε, η ομάδα Μίνσκ, όπου συμμετέχει η Ρωσία ως μέλος. Όπως ε, σε είπα, πήγα τον περασμένο μήνα στο Νότιο Κάφκασο και ανησυχούμε για την έλλειψη προόδου σε αυτές τις συνομιλίες. Η ένταση είναι πάρα πολύ αισθητή στην περιοχή. Και επίσης η Ρωσία θα πρέπει για τη Γεωργία να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου 2008. Ολοκληρώνοντα, βλέπουμε ότι έχουμε πολλά θέματα με τη Ρωσία που αφορούν την οικονομία, την κοινωνία μας και τις στρατηγικές μας ανησυχίε. Ε, έρουμε τους φραγμούς στο εμπόριο, στη μετακίνηση και στην ανταλλαγή και περιμένουμε ε, να έχουμε όλο και περισσότερη σύγκληση και επαφές των πολιτών. Φιλοδοξία μας είναι οι σχέσεις μας με τη Ρωσία να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για τη διαδικασία εξυγχρονισμού που θα πρέπει πάντα να είναι και οικονομική αλλά και πολιτική και το τονίζω αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπέτε πρόσωπε. Εκ μέρου των ομάδων τώρα από το και δύο λεπτό. ο κύριο Κέλαμ. Ευχαριστώ. Κυρία Υπέτη εκπρόσωπε, νομίζω ότι η σημερινή στιγμή είναι πολύ σημαντική λίγο πριν την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας γιατί υπήρξε τι αλλαγή συμπεριφοράς αλλά και ε, γενικώ ψυχικής κατάστασης των Ρώσων πολιτών. Γιατί φαίνεται ότι συντελείται μια αλλαγή της νοοτροπίας ε, εκ μέρου των Ρώσων πολιτών που έχασαν πια την αδιαφορία τους για τα πολιτικά, λαμβάνουν ενεργό μέρος στην πολιτική ζωή και αυτό το είδαμε στις πρόσφατες εκλογές. Και δεύτερο σημείο είναι ότι το κόμμα του κυρίου Πούτιν πέρασε στη μειοψηφία. Σε συνάντηση της περασμένης εβδομάδας στις Βρυξέλλες με τον κύριο Κασπάροφ και τους ηγέτες της ρωσικής αντιπολίτευσης έδειξε ότι το 49% δεν είναι το πραγματικό αποτέλεσμα. Το πραγματικό αποτέλεσμα για τον Πούτιν είναι γύρω στο 30%. Οπότε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε στις αλλαγές και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία. Το να κάνουμε σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα δεν αρκεί. Όπως είπε η κυρία Σαρτσόβα, ε, μέχρι στιγμής η Ρωσία υποκρινόταν ότι έχει δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποκρινόταν ότι πιστεύει τη Ρωσία. Αλλά έχει περάσει πια αυτός ο καιρός και θα πρέπει να αντιδράσουμε και απέναντι στη Ρωσία όπως αντιδράσαμε και απέναντι στην Αραβική Άνοιξη γιατί μπορεί να λάβει χώρα μια Ρωσική Άνοιξη και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Σας ζητώ λοιπόν κυρία Υπατή εκπρόσωπο να διαμηνήσετε αυτή τη σκέψη προς τους ομολόγους μας της Ρωσίας ότι λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά τις προθέσεις και την ετοιμιγορία των Ρώσων πολιτών και ότι οι ηγέτες της Ρωσίας θα πρέπει να αλλάξουν το ύφος και το στυλ τους. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και κάποιους περιορισμούς ε, προς αξιωματούχους που ασχολούνται με την έκθεση Μακμπίση και με τις εκλογές. Ευχαριστούμε κυρία Κέραν. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Φόμποντα. Κύριε Ήπατη εκπρόσωπε, νομίζω ότι επίκειται μια πολύ σημαντική συνάντηση κορυφής για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω του διαλόγου που πρέπει να έχουμε με την ηγεσία της Ρωσίας. Αναφέρομαι στον ενεργειακό διάλογο, ε, στην ολοκλήρωση της ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ ε, και έχουμε και μια συμφωνία συνεργασίας επί της οποίας πρέπει να εργαστούμε. Και ελπίζω να ε, ξαναξεκινήσει το θέμα. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα των εκλογών όπως ε, το θίξατε κι εσείς και άλλοι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξεκάθαρη θέση σας, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε. Νομίζω ότι είναι δείγμα οριμότητας εκ μέρους ε, των πολιτών της ε, Ρουσίας το γεγονός ότι δεν αποδέχονται οτιδήποτε προέρχεται από το Κρεμλίνο, από τον ρωσικό λευκό οίκο. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, η οποία προσπαθεί να πείσει το πολιτικό κατεστημένο ότι είναι καλύτερα να ακολουθήσουν άλλο δρόμο, δημοκρατικό, ανοιχτό. Αυτή η γραμμή πρέπει να επιβληθεί. Έχουμε λοιπόν το κοινό μας ψήφισμα όπου αναφέρεται, όπως είπατε και εσείς, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, ότι πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή που είσαι ο κ. Μεντβέντεφ να εξετάσει το θέμα με ειλικρίνεια. Μαζί με τον κύριο Φλάκενστάιν πήγαμε στη Ρωσία στις αρχές Νοεμβρίου και ήδη τότε διαπιστώσαμε ότι θα υπήρχαν σημαντικά προβλήματα στις ε, εκλογές ε, και ελπίζουμε αυτή η έρευνα να παρουσιάσει χρήσιμα αποτελέσματα. Ε, πρότεινα να οργανωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ακρόαση ε, τον Ιανουάριο με τα κόμματα που συμμετείχαν, με αυτά που δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν ε, με τον ΟΣΑ, με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, να αποκτήσουμε μία σφαιρική εικόνα. Τώρα λοιπόν θέλω να απευθύνουμε έκκληση στο κοινό μας ψήφισμα ε, σχετικά με την επανάληψη των εκλογών. Ας περιμένουμε λιγάκι, ας δούμε τις λεπτομέρειες, τα γεγονότα. Ίσως να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα ότι πράγματι, ίσως καταλήξει και ο Μεντιέντεφ στο αποτέλεσμα, στο συμπέρασμα, ότι σε ορισμένες εκλογές πρέπει να επαναληφθούν, σε ορισμένες περιοχές πρέπει να επαναληφθούν εκλογές. Αλλά καλύτερα να περιμένουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο κυρία Όγιουλαν για δύο λεπτά επίσης. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, το πρωταρχικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ε, Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι η νομοποίηση ε, της ε, Ντούμα μετά τις πρόσφατες εκλογές. Λαμβάνοντας υπόψη τα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα διεθνών οργανώσεων παρατήρηση εκλογών, η νομοποίηση της εκλεγής σας Δούμας είναι συζητήσιμη. Ε, φαίνεται ότι υπήρξαν πολλές ε, ατασταλίες ε, στις εκλογές και δεν επιτράπηκε εγγραφή σε ορισμένα κόμματα. Κάτι που καταστρατηγεί το νόμιμο δικαίωμα των ε, Ρώσων πολιτών να εκλέξουν τους εκπροσώπους στους ελεύθερες και ανώθευτες εκλογές. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι οι υποσχέσεις του Πρόεδρου Μετβέντεφ να ελέγξει τα αποτελέσματα ε, των εκλογών είναι ε, έγκυρες. Παρόλο που η Ρωσία εξακολουθεί να είναι σημαντικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οικονομικό μας συμφέρον θα πρέπει να επισκιάσει τις αρχές της δημοκρατίας που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες της. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά πώς θα προχωρήσει απέναντι σε μια κυβέρνηση που στερείται νομοποίηση για να εκπροσωπεί τους πολίτες. Ε, δεν θα πρέπει να ανεχτούμε το αυταρχικό καθεστώς του Πούτιν. Δεν θα πρέπει το Κρεμλίνο να μετατρέψει τη Ρωσία σε, σε απολυταρχικό κράτος. Η ομοία αλήθεια λέει ότι με τον Πούτιν και τους ε, στο Κρεμλίνο δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους ε, στόχους μας ε, ως προς τη Ρωσία. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει οι ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές που έχουν συλλάβει και επίσης οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις, ιδιαίτερα αυτές που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ευρώπης στην ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ρωσία θα πρέπει να διεξαγάγει νέες ελεύθερες και ανώθευτες εκλογές. Για δύο λεπτά το λόγο ο κύριος Σούλτς. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, η συνάντηση Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία λαμβάνει χώρα αυτήν την εβδομάδα με σούση ε, μια ε, πολύ τεταμένη κατάσταση. Οι προσπάσει εξυγχρονισμού ε, των τέρνων μα θα κριθούν από το κατά πόσον ε, θα υπάρξει πράγματι εξυγχρονισμός τη κοινωνία με περισσότερη δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την έκθεση της ΟΝΤΙΡ ε, και από τον, ε, τους ελέγχους που έχουν γίνει προέκυψε ότι η Δούμα ποδηγετήθηκε και υπήρξαν διαβλητέ εκλογές. Η Στη Ρωσία δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία. Διαμαρτυρήθηκαν 10.000 άνθρωποι, αυτοί αισθάνονται εξαπατημένοι και θεωρούν ότι πιστεύουν ότι προσβλήθηκαν, ε, δεν επιτράπει να συμμετάσχουν πραγματικά ακόμα τα αντιπολίτευση. Ακόμα και ο Κορμπατσόφ μέχρι τώρα δεν επέκρινε τον Πούτιν. Ο Κορμπατσόφ ζητάει τώρα ε, νέε εκλογέ και την ακύρωση αυτών που έλαβαν χώρα. Εμεί δεν πρέπει απλά να παρακολουθούμε κατά πόσο η Ρωσία θα τα καταφέρει μόνη τη ε, να πετύχει. Γιατί φαίνεται ότι πια είναι μια νέα εποχή. Είναι αστείο να περιμένουμε από εκείνου ανεξάρτητη έρευνα ε, τη στιγμή που φέρουν την ευθύνη. Και στη τελική ανάλυση τι περιμένουμε από ένα πρόεδρο Μεντιέντεφ, ο οποίος επί τέσσερα χρόνια ήταν αντιπρόεδρο αντιπρόεδρος ε, υπό τον Πούτιν. Υποτίθεται αυτό θα τα ελέγξει και υποτίθεται ότι ξέρει ότι δεν συνέβη τίποτα το μεμτό. Και μάλιστα όμως ε, απειλεί εκείνου που υπέβαλαν διαφορετικού αριθμού. Ο Μεντιέντεφ έχει την δυνατότητα να αποκαταστήσει όλες τις φρούδες ελπίδε είχαν συνδεθεί με το όνομά του και αυτό θα το κάνει μόνο αν προκηρύξει νέε εκλογέ. Και αυτό ο Πούτιν που έβγαλε από την τσέπη του το όπλο τη Καγκεπέ, τι περιμένουμε από ένα στιγνό εγκληματία, ο οποίο εδώ και χρόνια ε, ποδοπατά τι κραυγέ ε, τη κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει με τον συνηθισμένο τρόπο να ζητήσει απλά έρευνες από τη ρωσική πλευρά τη στιγμή που οι νέε διαφανεί εκλογέ. θα ήταν το σωστότερο, όπω επίση και το να επιτραπούν ε, τα απαγορευμένα κόμματα. Γι' αυτό λοιπόν σα παρακαλώ αύριο να στηρίξετε τη δική μα την τροπολογία. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο Μιγκάλσκι. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άστον για το, την υπενθύμηση που μας έκανε ότι η Ρωσία ε, δεσμεύεται από την κατάσταση ε, των από την υπόσχεση να τηρήσει το σχέδιο των έξι σημείων του Σαρκόζη για τη Γεωργία. Χαίρομαι που το υπενθυμίσατε την υποχρέωση αυτή τη Ρωσία. Επίση, σε ό,τι αφορά την αντίσταση ή την διαφωνία σε ό,τι αφορά τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα των τελευταίων εκλογών και την στήριξη της Αφύπνιση τη ρωσική κοινωνία. Υπάρχει φαίνεται πολιτική βούληση. Φάνηκε από αυτά που είπαν ο κύριος Κέλαμα από το ε, ΕΛΚΟ, ο κύριος Σβόμποντα, ο κύριος Σούλτ και το δικό μας κόμμα, οι συντηρητικοί και οι μεταρρυθμιστές ε, είναι αποφασισμένοι ως προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στην αφύπνιση της ρωσικής κοινωνίας και να στηρίξουμε αυτή την κατάσταση και μόνο υπό αυτό τον όρο θα γίνει πραγματικά αυτό που επιθυμούμε η Ρωσία, δηλαδή ένα σημαντικός οικονομικός μας εταίρος αλλά και σημαντικός πολιτικός εταίρος. Γι' αυτό και σα ενθαρρύνω κυρία Άστον και βλέπετε ότι στο θέμα αυτό τη χάνετε τη υποστήριξη υποστήριξης σα σύσσωμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστούμε κύριε Μιγκάλσκι για ένα λεπτό το λόγο κύριο Σόλτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αστόν, τα στρατηγικά συμφέροντα ε, θα πρέπει να συνδυάζονται με τις ε, επιθυμίε των ε, πολιτών να αντιμετωπιστούν οι κοινέ προκλήσεις. Στρατηγικό σημαίνει παράλληλα ότι θα πρέπει να προβληθεί το κοινό. Στρατηγικό όμως σημαίνει ότι διεκδικεί κανείς το συγκεκριμένο, το να είναι οι διαδικασίες, οι πολιτικές διαφανείς για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών. Μεταξύ μας συμφωνούμε. Τίποτα δεν δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Εκείνο όμω που δεν κατανοούμε είναι γιατί η κοινή ασφάλεια δεν μπορεί να ε, υλοποιηθεί με κοινό τρόπο. Έχουν κατατεθεί προτάσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επόμενη συνάντηση κορφή πρέπει να λάβει υπόψη τη αυτέ τι ε, προτάσει. Ε, θα πρέπει τα κονδύλια να συμπεριληφθούν αντί για εξοπλισμού σε εξυγχρονισμό τη κοινωνία. Γιατί αυτό θα ωφελήσει και τι δύο πλευρέ και του πολίτε οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και αυτοί δικαίω ε, στην ευημερία. Οι ευημερούσε ε, κοινωνίες σε τελική ανάλυση ε, σέβονται την εξουσία γιατί κοινωνίες ευημερούσες χρειάζονται τη στράτευση όλων των πολιτών. Οι διαδηλωτές στη Ρωσία επισήμαναν όλα αυτά τα γεγονότα στην εξουσία και ζήτησαν, υπέβαλαν συγκεκριμένα αιτήματα. Ο κύριος Μπέλτε. Για ένα λεπτό και επιμένω λίγο γιατί πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προειδοποίηση γρήπη εξέδωσε η ύπατη αρχή δημόσια υγεία και ο εκπρόσωπο Γεννάδη Νιτσέγκο στι 10 Δεκεμβρίου, μέρα Σάββατο, αλλά δεν ευδοκίμησε αυτό. Δεκάδε χιλιάδε πολιτών παρόλα αυτά ε, διαδήλωσαν για τις προφανείς νοθείες των ε, εκλογών στις 4 Δεκεμβρίου. Ήταν πολιτική ε, μανούβρα και λιγμός ε, αυτός του Νισέγκο και ο κόσμος ε, αντί να υποκύψει διαδήλωσε κατά της άρρωστης κοινωνίας και ενός συστήματος και δίκαια. Είναι πραγματικά ανάγκη να γίνει μια αυτοκριτική και από πλευρά των Ρώσων, ιδιαίτερα ενώπιση των προεδρικών εκλογών το Μάρτιο του 2012 θα συζητήσετε τα εσωτερικά, αλλά παρακαλώ να συζητήσετε και ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής. Πώς εκτιμάτε ε, τις πιθανότητες να είναι πιο θετική ε, η Ρωσία απέναντι στη Δύση σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ε, πώς μπορούμε να λύσουμε με ειρηνικό τρόπο αυτή την έφλεκτη υπόθεση. Ελπίζω αυτό να είναι πρώτη προτεραιότητά σας όταν συζητάτε ε, με το Ιδιανδρία Πούτιν και με Τβιέντεφ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Όμεν για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, αυτή η σύνοδος κορυφής έχει να κάνει με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα είναι ε, να ενισχύσουμε, λέτε, τους δεσμούς μας με τη Ρωσία. Μου επιτρέπετε να σας πω, Πρόεδρε, ότι ε, από αυτή την άποψη μπορεί να είναι θετική η έκβαση. Ε, διότι θα μπει στον ΠΟΕ η Ρωσία και αυτό σημαίνει επίσης ότι θα υπάρχει και μια δυνατότητα επιτάχυσης των διαδικασιών για την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Και αυτό το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ενέργεια, διευκόλυνση θεωρήσεων διαβατηρίων, επενδύσεις ε, κατέρωθεν των επιχειρήσεων, χωρίς διακρίσεις, χωρίς προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε επιγόντως. Αλλά, πρόεδρε, υπάρχει και το αλλά. Σε μια εταιρική σχέση ανήκουν και αξίες και γνήσιες αξίες. Το είπατε και εσείς, κυρία, είπατε εκπρόσωπε. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αξίες για μας και η Ρωσία έδειξε ότι στις εκλογές για τη Δούμα δεν σέβεται τέτοια πράγματα. Έλειψε ο σεβασμός από τις εκλογές. Πρόεδρε, σε ορισμένες ε, ε, ε, περιφέρειες κάποια κόμματα έφτασαν και το 100% των ψήφων. Μάλιστα, έχουν και πρόβλημα στην αριθμητική σήμερα, περισσότερο από τους πρώην Ούτε τα μαθηματικά δεν σέβονται, 100%. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να αποτραπεί να ε, ζήσουμε το ίδιο δράμα και την ίδια καταπάτηση των αξιών και των ελευθέρων εκλογών που ζήσαμε και τώρα. Συμφωνήστε το με τον κύριο Μετβέντεφ να λυθούν αυτά τα πράγματα. Έτσι και με έναν τρόπο λίγο στεναρό. Πρόεδρε, μια χώρα που επικαλείται αυτές τις αξίες πρέπει να ξέρει ότι μία από τις βασικές αξίες είναι η δημοκρατία και ότι εκλέγεσαι ε, με δημοκρατικές διαδικασίες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Φλέκενστάιν για δύο λεπτά. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Άστον, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η κυρία Όμεν Ρόιτεν σχετικά με τις εκλογές και η θερμή μας παράκληση απευθύνεται στον Ρώσο Πρόεδρο να του καταστήσουμε σαφές ότι μετά από τις δηλώσεις του θέλουμε να δούμε πράξεις και θα ελέγξουμε ακριβώς αυτά που είπε. Σωστά είπε ο κύριος Σφόμποντα να διοργανωθεί μια μεγάλη ακρόαση όταν θα έχει καταθέσει την πρότασή της η ΟΝΤΙΡ και θα θεωρούσα λάθος πριν υπάρχει έκθεση αυτή να ζητήσουμε επανάληψη των εκλογών. Ο κύριος Κέλαμ δεν είναι πια εδώ, αλλά θα ήθελα να πω στον κύριο Κέλαμ, ίσως να ήταν ε, και λάθος ε, μετάφρασης, να του πω ότι οι διαδηλωτές στη Μόσχα αποτελούν ευκαιρία και για μας. Όμως αυτό είναι λάθος. Δεν είναι ευκαιρία για μας, είναι ευκαιρία για τους ίδιους τους ανθρώπους στη Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα έπρεπε να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτά που λέμε. Οι εκλογές είναι σημαντικό θέμα στη συνάντηση κορυφή, αλλά αυτή η συνάντηση κορυφής μπορεί να εξελιχθεί και σε ε, συνάντηση αισιοδοξία. Δύο πράγματα θέλω να πω. Μετά από 18 χρόνια διαπραγματεύσει ένταξη στον ΠΟΕ. Και έτσι θα ξεκαθαριστούν οι κανόνε του παιχνιδιού και θα διευκολυνθεί η συμφωνία με εμά. Μονομερεί ε, περιορισμοί εμπορικοί, όπως υπήρξαν, ελπίζουμε στο μέλλον να μην επαναληφθούν. Και ε, η επιβάρυνση, όλα αυτά επιβάρυναν τις, ε, τα δικαιώματα υπερπτήσεων στη Σιβηρία. Κάτι άλλο για τις ε, θεωρήσεις και για την κινητικότητα. Χαιρόμαστε που θα υπάρξει μια ρύθμιση ε, σχετικά με τις, τη σύνδεση της μεταφορές στο Καλίνιγκρατ. Αυτό είναι μεγάλη διευκόλυνση για τους Ρώσους αλλά κυρίως για το Καλίνιγκρατ. τα κοινά βήματα ελπίζουμε αν υπάρχει καλή θέληση και των δύο κρατών θα οδηγήσουν κάποια στιγμή να εφαρμοστεί αυτό το καθεστώ απαλλαγή από θεώρηση. Μιλάμε για εξυγχρονισμό, για ανθρώπινα δικαιώματα, για οικοδόμηση τη κοινωνία των πολιτών. Ε, θέλουμε όλα αυτά να καταλήξουν σε αίσιο τέλο, αλλά αν δεν υπάρχει η ανθρώπινη επαφή, όλα αυτά δεν αξίζουν τίποτα. Ε, μπλε κάρτα από τον κύριο Μιγκάλσκι, τη δέχεστε, όχι, όχι, δεν τη δέχομαι. Καλώς. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Πόσελτ για 1,5 λεπτά. Frau Präsidentin, sehr geehrte Lady Ashton. Ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Lady Ashton. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Πουτίν δεν είναι μόνο αντιδημοκράτης, είναι αντιδημοκράτης μεγάλου βεληνικούς. Ας μην ξεχνάμε πως ανέβηκε στην εξουσία, κέρδισε τις εκλογές ε, εξαπολύοντας ε, όλητρο κατά της ε, Τσετσενίας. Και σε όλη του τη θητεία και ως ε, πρόεδρος και ως υπουργός εξωτερικών δεν έκανε τίποτα άλλο από το να οδηγήσει την Ρωσία στην οπισθοχώρηση, στην καθυστέρηση σε όλους τους τομείς. Και ο κύριος Μεντιέντεφ ναι να έχει ένα πιο συμπαθητικό πρόσωπο αλλά στην, Ιερά, στην Αγία Γραφή αναφέρεται να τους κρίνεται από τα αποτελέσματα. Και εμείς δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι αιτιολογημένο το αίτημα στη Ρωσία να υπάρξουν δημοκρατικές εκλογές. Μα δεν έχει νόημα ε, το να παρακαλούμε εκείνους ε, που χειραγώγησαν τις εκλογές να ελέγξουν και να αποκαλύψουν ε, αυτή τους την πράξη και ακούμε ότι αυτό που προέχει στη Ρωσία είναι σταθερότητα. Αυτό ε, το ε, είπαμε και για την Αφρική ε, και στην αρχή είχαμε κροκοδίλια δάκρυα για τον Καντάφη, τον Μουμπάρακ. Όσον αφορά τη Ρωσία μας ενδιαφέρει η σταθερότητα. Όμως σταθερότητα μπορεί να υπάρξει μόνο αν στη Ρωσία έχουμε δημοκρατικό κράτος δικαίου όπως ακριβώς το εκπροσωπούν οι διαδηλωτές στη Ρωσία για την δημοκρατία και την ελευθερία. Σταθερότητα χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι ένα δίδαγμα που επιτέλους πρέπει να εξάγουμε από την ιστορία. Σας ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Βιγγένιν για ένα λεπτό. Κυρία Άστον, θα ήθελα ε, σε αυτή αυτή τη στιγμή να σας επιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέματα. Φαίνεται ότι ε, χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία για να κάνουμε γενικές αξιολογήσεις για όλες τις τυχές της ζωής της Ρωσίας. Αυτό βέβαια δεν βοηθάει και πολύ γιατί χάνουμε αποσπάτη προσοχή μας. Αυτή τη φορά δεν χάσαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκτίμηση και να υποβάλουμε και κάποιες συστάσεις ό,τι αφορά το πρόβλημα των εκλογών της Ρωσίας, ευελπιστώντα ότι οι προεδρικές εκλογές του χρόνου θα είναι καλύτερα προετοιμασμένε, ε, θα τύχουν σωστότερη διαχείριση και θα είναι πιο ελεύθερες και πιο δίκαιες. Παρά τις επικρίσεις μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι η Ρωσία σήμερα είναι διαφορετική και θα πρέπει αυτή την ε, θετική στιγμή να την αξιοποιήσουμε όχι μόνο για να κατηγορούμε τις αρχές αλλά και να τους αθαρρύνουμε να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους ώστε να αισθανθούν την υποστήριξή μας και αυτοί που δίνουν μάχη υπέρ της δημοκρατίας στη Ρωσία. Θα πρέπει επίσης ε, να ζητήσουμε τη συνεργασία της Ρωσίας για να εξασφαλίσουμε ε, σταθερότητα, υφόρο οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ανάπτυξη στην περιοχή της γειτονίας μας. Και η νέα ηγεσία που θα διαμορφωθεί στη Ρωσία του χρόνου δεν θα πρέπει να εμπλακεί σε ανταγωνιστικές διαμάχες, αλλά να βοηθήσει στην απεμπλοκή ιδιαίτερα των παγωμένων συγκρούσεων στον Κόρνο Καραμπάχ και την υπερδινιστερία. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye και πρώτα θα ακούσουμε για ένα λεπτό την κυρία Αντρικένα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Κασιάνο, τον πρώην Πρωθυπουργό που παρακολουθεί τη συζήτηση. Ε, κάποια σημεία που δεν περιλαμβάνονται στο ψήφισμα. Ε, ο Μετβέντεφ, ο Πούτιν και το κόμμα τους έχασαν τις εκλογές στη Δούμα. Δεν έχασαν μόνο ε, πολλές στη Δούμα, αλλά έχασαν ουσιαστικά τις ίδιες εκλογές. Ήταν φανείς οι παραβιάσεις των εκλογικών διατάξεων και η νοθεία στον, στις εκλογές. Έγινε, υπήρξαν τα και στην καταμέτρηση των ψήφων. σίγουρα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να αξιολογήσουμε ως δίκες τις εκλογές στη Ρωσία. Φαίνεται ότι καταστρατηγήθηκαν τα εκλογικά δικαιώματα των Ρώσων πολιτών. Ο Μιχαήλ Κορμπατζόφ, ο πρώτος και τελευταίος πρόεδρος ε, της ε, Σοβιετικής Ένωσης ε, αναγνώρισε αυτές τις τασέλειες και ζήτησε να διεξαχθούν νέες εκλογές. Δεν θα πρέπει να το παραγνωρίσουμε λοιπόν αυτό. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, α, διακόπηκε δυστυχώς η κυρία Δρικένε. Ο κύριος Ταμπάιτζ. Ευχαριστώ ως παρατηρητής των εκλογών μετέβη στη Ρωσία και διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε δίκαιος πολιτικός ανταγωνισμός, δεν υπήρξαν ίσες ευκαιρίες μεταξύ των διαφόρων πολιτικών κομμάτων ε, και το θέμα του εκλογικού νόμου ε, είχε κάποια προβλήματα και η πρόσβαση των κομμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν προβληματική και ούτω καθεξής. Πάντως ήταν λάθος εκ μέρους μας να ζητήσουμε διεξαγωγή νέων εκλογών στη Ρωσία. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος ε, να συμπεριφερθούμε στη Ρωσία. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι η συνεργασία με τη χώρα αυτή. Φυσικά θέλουμε ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές, αλλά διαφωνώ με προλαλήσαντες. Σίγουρα η Ενωμένη ε, Ρωσία έχασε την πλειοψηφία, υπέστη σημαντική ε, σημαντικό πλήγμα στις εκλογές ε, το κόμμα του Πούτιν, αλλά παρόλα αυτά η δημοκρατία σημείωσε πρόοδο στη Ρωσία. Και μάλιστα σήμερα υπάρχει ε, ισχυρή αντιπολίτευση και στη Δούμα και στο Ρωσικό Κοινοβούλιο, αλλά και διαμαρτυρίες στους δρόμους. Έδειξε ε, οι διαδηλωτές τη διαφωνία τους με το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο κύριος Ιβο Βάγγελ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λέει Άστον, είπατε εκπρόσωπε, επιτρέψτε μου καταρχάς να καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν εξέχοντα προσκεκλημένο μας που έχει και μεγάλες προσδοκίες, τον κύριο Μιχαήλ Κασιάνοφ που παρευρίσκεται στο θεωρείο. Νομίζω άνθρωποι σαν τον κύριο Κασιάνοφ αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες για το θάρρος τους και δεν θα πρέπει να τους παραβλέπουμε και να τους λησπονούμε σε επαφές μας με την επίσημη ηγεσία της χώρας. Στο παρελθόν είχαμε πολλές διαπραγματεύσεις και συνομιλίες με την κυβέρνηση της Ρωσίας και παραλείψαμε να ασχοληθούμε με την αντιπολίτευση. Ελπίζω, λέει Κάσια ε, Άστον, να ε, τους διαβιβάσετε ότι περιμένουμε περισσότερα ε, από τη Ρωσία και για το ε, Ορεινό Καραμπάχ και για άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βάγκρο. Δόκτωρ Τάνοκ. Πρόεδρε, οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία έδειξαν ότι έχει επιδεινωθεί η δημοκρατία στη χώρα. Εκτεταμένη νοθεία, παρενόχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, ειρηνικών διαδηλωτών, ε, όλα αυτά ε, διαψεύδουν τον κύριο Πούτιν ότι ήταν ελεύθερες και δίκαιες οι εκλογές. Ακόμα και το βασικό κόμμα τη αντιπολίτευση το ΠΑΝΑΣ, κόμμα τη ελευθερία ΛΟ, δεν είχε δικαίωμα να καταγραφεί και να συμμετέχει σε εκλογέ. Θα πρέπει να θυμίσουμε στη Ρωσία ότι ω μέλο του ΟΑΣΕ και Συμβουλίου τη Ευρώπη είναι υποχρεωμένο να ε, διαφυλάσει την αστηριότητα και την ακαιρεότητα των εκλογών. Θα πρέπει να σταματήσει η μαζική διαφθορά και ο μαζικό πλουτισμό κάποιων υψηλών στελεχών, Όπω έδειξε η τραγική περίπτωση του Σεργέη Μαγνίσκη, που επέλεξε να καταγγείλει τη μεγαλύτερη περίπτωση φοροδιαφυγής και τον φυλάκισαν που έχασαν τη ζωή του μάλιστα στη φυλακή. Κύριος Μέλτσα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορεί να έχουμε 10.000 δυσαρεστημένους Ρώσους που έδισαν ένα μήνυμα. Κανείς όμως δεν έχει την ψευδέστηση ότι έρχεται αρκετή δύναμη για να κλονίσει το σύστημα αυτή η διαμαρτυρία για να αλλάξει εξουσία οι πολιτικές απόψεις των διαδηλωτών ε, είναι ετερόκλητες και ο ο Πούτιν ω σταθεροποιητή μετά το χάος ε, της δεκαετίας του 90 ε, χαίρει ακόμα μεγάλη εκτίμηση και υποστήριξη από την κοινή γνώμη που δεν θα πρέπει να την υποτιμούμε και από την οικονομία. Τέλος, η Ρωσία ως προς τις δημοκρατικές προδιαγραφές δεν μπορεί να μετρηθεί παρά μόνο περιορισμένα με ευρωπαϊκή είναι ακόμα στα, σπάρναγα, ε, σπάργανα ε, η ε, δημοκρατία και θα πρέπει να ξεπεραστεί η κληρονομιά 70 ετών κομμουνισμού. Θα πρέπει να προληφθούν στο μέλλον τέτοιες εξελίξεις, να προωθήσουμε τον εκδημοκρατισμό και αυτό θα πρέπει να το πει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο Κορυφής. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ αυτός ο γύρος ομιλητών με την κυρία Σενκλέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Άστον, χρειάστηκε να βγω λίγο στο τέλος προηγούμενης συζήτησης να απαντήσω σε ένα τηλεφώνημα ενός ψηφοφόρου. Συγγνώμη που θεωρείτε τόσο σημαντικό να είναι τα μέλη εδώ να σας ακούνε. Γεμάτο το κοινοβούλιο, 23 βουλευτές σας ακούνε. Κρίμα. Ήθελα να πω κάτι για τη Ρωσία όμως που είναι σοβαρή κατάσταση. Αλλά αυτό δεν δείχνει τους περιορισμούς που έχουμε. Η Ρωσία, η μεγάλη οργισμένη αρκούδα που προσπαθούμε να τη συνετίσουμε και να τη μάθουμε τρόπους. Έτσι δεν θα φτάσει ποτέ σε κανένα επίπεδο δημοκρατικής λογοδοσίας. Αλλά εσείς πού να ξέρετε από τέτοια πράγματα. Ξέρετε ότι οι Ρώσοι ονομάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση παροδικό φαινόμενο. Ελπίζω να έχουν και δίκιο κατά τα άλλα. Μπορούμε να συζητούμε μαζί μας, αλλά αυτοί θα κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό δείχνει πόσο περιορισμένοι είστε εσείς στη δράση σας. Με την παρέμβαση κυρίας Ινκλέρ ολοκληρώθηκε ο γύρος των ομιλητών που ζητούν αυθόρμητα το λόγο και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Άστον για να ολοκληρώσει και να απαντήσει σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν στη συζήτηση. Αγαπητή Κάθριν, Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και να σας πω ότι τα μηνύματα που στείλατε ήταν ιδιαίτερα ευκρινή και ε, θα τα διαβιβάσω. Ε, πράγματι θα τεθεί το θέμα των εκλογών, αυτό είναι σαφές και θέλω να πω στον κύριο Κάλαμ ότι παρακολουθούμε του σύνεγγυ στην ε, περίπτωση Μαγνίτσκι γιατί πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα όπως το είπε και ο ίδιος. Και εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ε, υπάρξει την Πέμπτη μία συνάντηση και με την κοινωνία των πολιτών, το φόρουμ το σχετικό στη Ρωσία. Θέλω να συζητήσω μαζί τους τα τελευταία γεγονότα και γενικότερα τη σχέση μας. Πάντα συζητάμε τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουμε στη συνάντηση κορυφή. Οι δικοί μου συνεργάτε ε, συναντήθηκαν με τον ε, πρώην Πρωθυπουργό ε, που είναι εδώ, το χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ και εγώ συναντήθηκα μαζί του τον Ιούλιο. Σε όλε τι συζητήσει με τη Ρωσία τίθενται μια σειρά θεμάτων, η γεωργία είναι ένα εξ αυτών. Σε συζητήσει για την εξωτερική πολιτική Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που και αυτά θίγονται. Για το Ιράν να έχετε δίκιο που το θίξετε το θέμα. Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ε, αφιερώνω πολύ χρόνο για να δω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Η Ρωσία είναι μέρος ε, του 3 συν 3, ε, συνεργάζεται με μας για να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να πείσουμε το Ιράν να μην ε, χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που ανησυχεί όλους. Όταν μιλάμε για την ε, κοινή γειτονία, όπως την αποκάλεσε ο Ξημότιβος Βουλευτής, συζητάμε τα θέματα της υπερδνηστερίας και του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και όπως είπα, είπα προηγουμένως στη συζήτησή μας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πρόοδος. Ε, όταν ήμουν στο Αζερβαϊτζάν και όταν επισκέφθηκα και την Αρμενία ανησύχησα με το πόσο τεταμένη είναι η κατάσταση. Η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει ε, να εξευρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. Νομίζω αυτά που ελέγχθησαν ε, δείχνουν ότι εμείς παίρνουμε τη δημοκρατία σοβαρά και περιμένουμε το ίδιο και από τη Ρωσία και τον κύριο Κλάμ, ε, κυρία Κλάμ, θέλω να πω, μάλλον δεν είναι πια εδώ, θέλω να της πω ότι αυτά τα οποία είπε δεν με προσέβαλαν δεν ε, πουδενή. Έχουμε λάβει έξι ε, προτάσεις ψηφίσματος για το θέμα αυτό. Μία από τους πράσινους, άλλη από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, τρίτη από τους φιλελεύθερους, από τους μεταρρυθμιστές